καταπολέσουμε τη βία και να εξασφαλίσουμε την ισότητα των φύλων. Περνάμε τώρα στο άρθρο 150, παρεμβάσεις διαρκείας ενός λεπτού. Κυρία Μπασέσκο, ένα λεπτό. προσπαθήσαμε να συμμετάσχουμε στο σύστημα αντιμετώπισης των πυλάβρων της ασπίδας κατά των πυράβλων. Αυτό έγινε πέρσι στις 8 Μαρτίου και προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε και εμείς. Θα έχουμε 8 επί 3 ασπίδες στην ε, Ρουμανία και αυτό από, τις, από το 2015. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το θέμα της αντιπυραυλικής άμυνας θα πρέπει να μας απασχολεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος διασποράς και διάδοσης πυρηνικών όπλων. Γίνεται λόγος για αντιμετώπιση της ε, κατάστασης έναντι ενδεχόμενου κινδύνου από τη ε, Ρωσία. Θα αρχίσουν όμως διμερείς ε, συναντήσεις για να φτάσουμε στη σύναψη συμφωνιών. Από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σας ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαστάμκος. Εκείνο από την μείζωνα παραδοχή ότι η εξυγίαση των δημοσίων οικονομικών ενός κράτους μέλους της Ευρωζώνης βαρύνει το ίδιο. Ωστόσο, απαιτείται συντονισμένη παρέμβαση για τη θωράκιση του κοινού νομίσματος έναντι των ε, κερδοσκοπικών παιγνίων αυτά που γίνονται τα κερδοσκοπικά παίγνια εις βάρος του ευρώ. η βαθύτατη δημοσιονομική κρίση στην ελλάδα αλλά και η δημοσιονομική ανισορροπία σε άλλα κράτη μέλη έφεραν στην επιφάνεια την ανάγκη συγκρότησης μιας πολιτικά κατευθυνόμενης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. με ερώτησή μου τη 17η Φεβρουαρίου 2010 προς την επιτροπή πρότεινα την καθίδρυση ενός ευρωπαϊκού νομισματικού ταμείου. με ικανοποίηση βλέπω ότι ο επίτροπος κύριος ρεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. περιμένουμε το ολοκληρωμένο σχέδιο εκ μέρους της επιτροπής. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ε, Σας ευχαριστώ κύριος Κάρλος Ευχαριστώ. Είδαμε ότι ο Ούγκο Τσάβες, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, συνεργάζεται με τρομοκράτες και δυστυχώς μπορούν να δράσουν στο έδαφος της Βενεζουέλας οι τρομοκράτες και βεβαίως κατέχουν και σημαντικές θέσεις. Δηλαδή, στην ουσία, ο Τσάβες συνεργάζεται με τους τρομοκράτες της ΕΤΑ ως Βάσκος θα ήθελα να στυλιτεύσω αυτή τη ε, στάση του στιγνού δικτάτορα Τσάβες και θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για να καταδικάσουμε τον Τσάβες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην ε, Προεδρία, δηλαδή στην κυβέρνηση του κυρίου Ροντρίγκε Θαπατέρο, ότι δεν θα πρέπει να δεχόμαστε με ανοιχτές αγκάλες ε, τρομοκράτες και αρχηγούς κρατών. Γιατί δεν μπορούμε να ταπεινωνόμαστε έναντι τους, ε, του Τσάβες όπως έγινε πρόσφατα. Διαφορετικά δεν καταδικάζουμε την τρομοκρατία όπως θα έπρεπε. Ε, Βασιλίκα Βορίκα Ταντσίλα. Η κυρία Βασίλη Βορίκα, Νταντσίλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ταμείο Αλληλεγγύης λειτουργεί καλά. Η κεκτηθήσα εμπειρία τα πρώτα χρόνια εφαρμογής μας καταδεικνύουν ότι υπάρχουν ε, κάποιες ανεπάρκειες στην εξέλιξη αυτού του Ταμείου. Δεν υπάρχει δηλαδή ταχύτητα απόκρισης ε, και διαφάνεια στη χρηματοδότηση αυτού του ταμείου, στη χρήση των κοντιλίων. Ε, αναφέρομαι ειδικότερα στις φυσικές καταστροφές. Σας υπενθυμίζω ότι η Ρουμανία υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τις πλημμύρες. Όμως τα χρήματα φτάσανε πολύ αργά σε σχέση με το σημείο το χρονικό στο οποίο θα ήταν αποτελεσματικά. Συνεπώς, Κάποιες προκαταβολές ίσως θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με μία πρώτη αξιολόγηση των ζημιών. Όταν έχουμε φυσική καταστροφή αυτό θα ήταν ένα πλεονέκτημα και οι πολίτες θα μπορούσαν να υποφοληθούν περισσότερο από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ο κύριος κοιτάντε τώρα. Για mucho tiempo que Fidel Castro ο Φιντέλ Κάστρο και η ολιγαρχία του έθεσαν τέλος στην επανάσταση της Κούβας. Κάτι το οποίο ήταν ολέθριο για όλους και ιδιαίτερα για την νεολαία ολόκληρου του κόσμου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την μεγάλη αυτή δικτατορία των αδελφών Κάστρο. Και αυτό που έχει σημασία είναι να θυμηθούμε και τον Φράγκο Ας μην ξεχνάμε τον και τον Φράνκο, ο οποίος ε, προσπαθούσε από το κρεβάτι του θανάτου να δικήσει τον κόσμο. Έτσι δρά και ο Κάστρο, όπως και ο Φράνκο. Θα πρέπει όμως να σώσουμε ζωές και να ε, μην θυσιάζουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Να διασφαλίσουμε δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού. Τάνια Φαϊρών. Παν Πάτ Δικόπ Cope Gallagher. Pan Gianni Presidente, Κύριε Πρόεδρε, ε, γνωρίζουμε ότι η Ισπανική Προεδρία επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις με χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής για συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ από τη διάσκεψη, διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής. Θα ήθελα να σας πω ότι επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις λησμονώντας σημαντικά θέματα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τήρησή τους. Στην Κολομβία συνεχίζονται οι δολοφονίες συνδικαλιστών καθημερινώς. Στην Ονδούρα επίσης υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία ε, κυβερνά μετά από ένα πραξικόπημα πέρσι και το ίδιο ισχύει και με τη Γουατεμάλα. Πρόκειται για πτυχές που αγνοούμε σκοπίμως. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή και η, και η Προεδρία να αντιμετωπίσουν πολύ σωστότερα το θέμα. Η κυρία Wallis, Diana Wallis. Μια και είναι η επέτειο τη μέρα των γυναικών αναφέρομαι σε ένα θέμα υγεία των γυναικών που εξακολουθεί να αφορά τι ταχτοπούδε. Πριν από δύο-τρία χρόνια ήμουν πάλι εδώ και μιλούσα για μια σιωπηρή και οδυνηρή ε, γυναική ασθένεια, την ενδομητρίωση. Καταστρέφει οικογένειες, ζωές και τη γονιμότητα. Ορισμένες γυναίκες δηλαδή δεν γίνονται ποτέ μητέρες. Και ίσως ε, επειδή έχει να κάνει με ε, γυναικολογικό θέμα. Ε, δεν θέλουμε να το συζητήσουμε. Ενδομητρίαση λοιπόν, έχει όνομα. Δεν είναι γνωστή ε, το αίτιο, δεν είναι γνωστό το αίτιο, δεν είναι γνωστή η αγωγή ε, και η αποθεραπεία. Λοιπόν, είναι η εβδομάδα συνειδητοποίηση του προβλήματος της στην Ευρώπη. Πότε θα σκεφτούμε σοβαρά αυτές τις γυναίκες. Επίτροπε, χαίρομαι που είστε εδώ και ελπίζω ότι θα δώσετε τα απαραίτητα κονδύλια σύντομα. Η κυρία Σαντρίν Μπελιέ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αναφερθήκατε στην καταιγίδα, την Ξύνθια, η οποία σκότωσε περίπου 60 ανθρώπους και έκανε μεγάλες ζημίες. Είναι μεγάλη λύπη αυτό αλλά είμαι και θυμωμένη σήμερα, διότι αυτή η ανθρώπινη καταστροφή θα μπορούσε να είχε αποφευθεί ή τουλάχιστον να έχουν μειωθεί οι επιπτώσεις της. Χθες στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη δημιουργούνται τεχνητές ακτές, παραβιάζοντας όλες τις νομοθεσίες. Η Natura 2000 και η προστασία αυτών των ζωνών είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε να μην έχουμε τέτοια φυσικά φαινόμενα στο μέλλον. Πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι στη διαχείριση. Πρέπει να εφαρμόζουμε αυστηρά το κοινοτικό δίκαιο και τις κοινοτικές ρυθμίσεις ε, για τα πτηνά, για τις ε, παραλίες κτλ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη βιοπικιλότητα. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μας φέρει σε μια νέα σχέση με τη φύση. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, την προηγούμενη εβδομάδα τα τσεχικά μέσα μίλησαν για το γεγονός ότι οι Γερμανοί πήραν πιο ε, αυστηρά μέτρα κατά οδηγών, τσέχων οδηγών από την άλλη πλευρά των συνόρων. Οι μάρτυρες λένε ότι έγιναν εξευτελιστικές εξετάσεις κατά των τσέχων. Δηλαδή υπέστησαν και ανάλυση ούρων. Οι Τσέχοι πολίτες μπορούν να κινούνται όπως θέλουν εντός της ζώνης ε, Σέγγεν και δεν πρέπει να υφίστανται τέτοια εξευτελιστική μεταχείριση. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διαβιβάσετε αυτά τα στοιχεία στις κατάλληλες αρχές έτσι ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα ε, μέτρα. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Κύριε Πρόεδρε, η Παγκόσμια ημέρα της ε, παχυσαρκίας θα πρέπει να μας απασχολήσει μέσα στα πλαίσια της συνδρομής ε, γιατρών και πολιτών για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Η 22η Μαΐου είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της παχυσαρκίας και έτσι θα προβάλλουμε μία ε, γενικότερη συνειδητοποίηση του προβλήματος ακούγοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Πρόκειται για ασθένεια και όχι πρόβλημα. Το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να υποστηρίξει αυτή την ε, πληθυσμιακή ομάδα. Οι στατιστικές παχυσαρκίας στην Ευρώπη ε, οδηγούν σε διαστάσεις καθαρής επιδημίας. Θα έχουμε 150 εκατομμύρια παχύσαρχους, δηλαδή 20% ε, του πληθυσμού και 15% του πληθυσμού θα είναι έφηβοι. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της ε, ε παχυσαρκίας. Ήλντα Φιγκεϊρέδο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επειδή μιλάμε για την εκατοστή επέτειο της ε, Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, θα πρέπει να δούμε και άλλα παράπλευρα ζητήματα, δηλαδή θέματα διάκρισης και κατά των γυναικών που, αποτελούν, που συνεχίζουν να αποτελούν θύματα ανισότητας. Θα πρέπει να τονίσουμε την επικαιρότητα αυτού του θέματος έτσι ώστε να υπάρχει ισότητα στον νόμο αλλά και στη ζωή. Βεβαίως ο ξέφρενος καπιταλισμός δεν βοήθησε την κατάσταση. Η επισφαλής εργασία, η φτώχεια, όλα αυτά αφορούν κυρίως τις, γυναίκες, τις γυναίκες που αποτελούν το 80% των φτωχών στην Ευρώπη. Οι γυναίκες δεν πρέπει να ξεχνάνε τα όνειρά τους. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις αδικίες και τις διακρίσεις προβάλλοντας νέους ορίζοντες για μια καλύτερη ζωή. Μπαύτον. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να να σας πω ότι πρόκειται να γίνει ένα δημοψήφισμα στην Ουαλία. Ναι, ένα δημοψήφισμα. Δεν μας δώσαν ένα για το Σύνταγμα, για τη Λισαβόνα, αλλά θα έχουμε για την Ουαλική Βουλή τώρα. Το θέμα είναι το εξής. Όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ουαλία, η Εργατική, το Λίπτεμς, και οι συντηρητικοί υποστηρίζουν αυτό το δημοψήφισμα και θέλουν ενίσχυση της Βουλής της Ουαλίας. Αλλά εγώ δεν θέλω. Μεταχειρίζονται άσχημα τους πολίτες και ε, αν περάσουμε και στην ανεξαρτησία στη συνέχεια θα έχουμε μεγάλες απειλές. Θα κλείσουν τα σχολεία, οι δρόμοι μας είναι χάλια και η πολιτική μας στο Κάρντιφ παρόλα αυτά θέλουν να προχωρήσουμε αυτή τη τρελή ιδέα της Βουλής της Ουαλίας. Δημοψήφισμα λοιπόν ελπίζω ότι θα καταψηφιστεί. Ο Πανμυρόσκαν Νικολάσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα συλληπιτήριά μας και να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με τα θύματα της Μαντέιρα. Η κατάσταση ε, απαιτεί γρήγορα μέτρα για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πέσαν τόσες πολλές ζημιές από τη φυσική καταστροφή. Ελπίζω ότι οι πορτογαλικές αρχές θα μπορέσουν να βοηθήσουν να προσδιορίσουν τις ζημίες και να βρουν και στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να τους στηρίξει. Τα χρήματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν για όσους επηρεάστηκαν από αυτή την καταστροφή. Ε, θέλω την υποστήριξή σας λοιπόν σε αυτό συνάδελφοι. Ε, υπάρχει και άλλη καταστροφή στην Αφρική, μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ κυρία Κολάσκα Βαβίνσκα. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Πρόσφατα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα για την Ουκρανία, στα πλαίσια τη οποία αναρωτιόμαστε αν ήταν σωστό να χορηγηθεί από τον τέος πρόεδρο τη Ουκρανίας ενό βραβείου στον Στέφαν Πρατέρα έναν ήρωα της, ε, της, του αγώνα για την εξαρτησία τη χώρα. Η παράγραφος αυτό οδήγησε σε πολλέ ε, κριτικέ στην Δυτική Ουκρανία. Θέλω να σας πω ότι αυτό το ψήφισμα δεν διαφυσβητούσε το ρόλο του Παντέρα για την εξαρτησία της Ουκρανίας του εναντίον τόνιζε την ανάγκη της αλεπερευθέρωσης της Ουκρανίας που στηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς. Αλλά το ψήφισμα αναφέρεται στο ότι ήταν λυπηρό που εδόθη το βραβείο αυτό χωρίς να ληφθούν υπόψη τα θλιβερά γεγονότα του πολέμου για την εξαρτησία της Ουκρανίας. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που έλειπε από το βραβείο που εδόθη στον Μπαντέρα ήταν μια έκφραση λύπης για τα θύματα, τα αθώα της, του αγώνα. Μόνο τότε θα μπορούσαμε να έχουμε πραγματικά αγώνα για την εξαρτησία της Ουκρανίας. Το βραβείο θα έπρεπε να συνοδεύεται από μια προσπάθεια συμφιλίωσης. Διακόπτει ο Πρόεδρος. A Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούστηκαν πολλές επικρίσεις ε, στο παρελθόν. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι υπάρχει η απόφαση της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το διατακτικό δεν μπορεί να συμβαστεί με τα βασικά δικαιώματα και τα εν λόγω έγγραφα του Συμβουλίου της Ευρώπης και επίσης με το Σλοβαγικό νόμο για την προστασία των μειονοτήτων. Αυτή η γνωμοδότηση ε, δεν αναφέρεται σε μια αναλογικότητα των μέσων και προβλέπει η ελεύθερη κυκλοφορία που είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εσωτερικής αγοράς να θεκυβεύεται αυτή τη στιγμή. Αυτή η νομοθεσία για την γλώσσα όπως έχει τροποποιηθεί είναι αντίθετη με διάφορες άλλες νομοθεσίες. Ιδίω όσον αφορά παραδείγματο χάρη το άρθρο 56 για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και επίσης το θέμα των οργάνων προσφοράς υγείας. Αυτή η διάκριση θα έλεγα ότι ακριβώς θα πρέπει να ε, δούμε ότι προστατεύει τα δικαιώματα όχι των πολιτών αλλά του κράτους και παρακαλούμε την Κομισιό να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε το κοινωτικό δίκαιο να εφαρμόζεται χωρίς περιορισμούς. Ευχαριστώ. Mulțumesc, domnule președinte. Θα σας μιλήσω για την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 30%. Το, τη δεκαετία του 80 φτάσανε στο 40% και συνέχεια στο 50%. Αυτά μας δίνουν τα στοιχεία της Eurostat. Δυστυχώς όμως έχει έχουν πληγεί οι τομείς όπου εργάζονται και άνδρας. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη διάκριση ανδρών και γυναικών και γι' αυτό στο νέο νομοθετικό πακέτο το οποίο θα προβάλλει η Κομισιόν θα πρέπει να υπάρχουν στόχοθετήσεις έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαφορές μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών και να μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας περισσότερο γυναίκες. Θα πρέπει δεν να ενταχθεί στο πακέτο Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. κύριε Πρόεδρε, Πρόσφατα γεγονότα στην Τουρκία επιβεβαιώσαν για άλλη μια φορά ότι τα δικαιώματα των συνδικάτων και των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, ε, καταπατούνται. Εδώ και μήνες, ε, δύο μήνες, 1.200 εργαζόμενοι του ΤΕΚΕΛ υποφέρουν από μαζικές απολύσεις και απώλεια των κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Κατά τη διάρκεια της απεργίας αυτής, ο πρόεδρος Ερτογάν ε, έχει απειλήσει να στείλει το στρατό για να αδειάσει το χώρο από τους ε, απεργούντες. Οι εργαζόμενοι ε, έχουν τύχει επίθεση από την αστυνομία με δακρυγόνα. Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να φροντίσετε στην Τουρκία να διχάνουν ισότιμες μεταχείρισης τα συνδικάτα και να εγγυούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα πρέπει να τηρούνται οι συμβάσεις ΙΛΟ. Ευχαριστώ. Κύριος Λουίτζιου Ντεμαγκίστρης. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά πρόσφατα στην Ιταλία είχαμε μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή στον ποταμό Πάδο. Δυστυχώς το ΔΕΚ μας καταδίκασε σε σχέση με την ρήψη απορριμμάτων και με τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα στην Καμπανία. Έχουμε μεγάλη αύξηση και λευκαιμίας, ιδιαίτερα στην ε, περιοχή του Κρότονα και του Τάραντο. Δυστυχώς ζούμε μια συνεχή περιβαλλοντική καταστροφή και θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει έτσι ώστε η Ιταλική κυβέρνηση να βρεθεί στο ύψος των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΔΕΚ μας καταδίκωσε για άλλη μια φορά τις προηγούμενες μέρες, διότι δεν μπορέσαμε να διαθέσουμε σωστά τα απορρίμματα. Και δυστυχώς επλήγει ιδιαίτερα η Νάπολη από αυτήν την κατάσταση. Πάνι Νικόλ Merci, Ευχαριστώ κύριε η συνδιάσκεψη του Λονδίνου για το Αφγανιστάν προκάλεσε πανικό στους Αφγανούς και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Το ειρηνευτικό σχέδιο που επικυρώθηκε από πολλές χώρες σημαίνει την ένταξη των Ταλιμπάν και πρέπει να γίνει μια μεγάλη συνέλευση σε ένα μήνα για αυτή τη συμφιλίωση. Οι γυναίκες δεν θέλουν, δεν πρέπει να πληρώσουν τη συμφιλίωση. Οι Ταλιμπάν θέλουν την κατάργηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την επιστροφή στη Σαρία. Και Υπάρχει ανησυχία, θα τραποποιηθεί το Σύνταγμα και θα καταργηθούν τα άρθρα που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των γυναικών. Ζητώ λοιπόν σήμερα επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθεί το μέλλον των γυναικών του Αφγανιστάν διότι δεν είναι δυνατόν να επανέλθουμε στο πιο γυναικοκτόνο καθεστώς που έχει δει πολύ ποτέ η ιστορία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουσουτήρα, ο επόμενος συμβιλτής. Σας ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι το ε, καθεστώς η διένεξη μεταξύ Λιβύης και Ελβετίας οδήγησε σε ολέθριες συνέπειες και αυτό αυτό αφορά εργαζόμενο στη Λιβύη και επενδυτές που δεν μπορούν να στείλουν, να αποστείλουν προσωπικό στη Λιβύη. Στο μεταξύ, εργαζόμενοι που βρίσκονται ήδη στη Λιβύη προσπαθούν να παραμείνουν ε, το περισσότερο δυνατόν, έτσι ώστε να βοηθήσουν όσους δεν μπορούν να προσέλθουν ή να επανέλθουν. Βεβαίως δεν ξέρουμε πόσο θα μπορέσει να διαρκέσει αυτή η κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όμοιρος μιας κατάστασης που αφορά δύο τρίτες χώρες. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει όλα τα μέτρα έτσι ώστε να επιληθεί το τρέχον ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε εξηγήσεις, επεξηγήσεις από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, διότι υποτίθεται ότι συνεργάστηκε με την ΕΤΑ. Και το Σάββατο είχαμε μια κοινή ανακοίνωση μεταξύ κυβέρνησης της Βενεζουέλας και της Ισπανίας σε σχέση με αυτό το γεγονός, επιβεβαιώνοντας αυτή τη συνεργασία Βενεζουέλας, Ισπανίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να μας χαροποιήσει ιδιαίτερα και να ε, εκφράσουμε την καλή μας θέληση προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, διότι θα πρέπει να καταπολεμήσει τη δράση της ΕΤΑ και δεν πρέπει να γίνεται χειραγώγηση ενός τέτοιου πολιτικού γεγονότος. Θα πρέπει να υπάρχει αυτόνομη δράση των δικαιοδοτικών και δικαστικών αρχών για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σμίτ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ισλανία ε, να πει κάτι για την συμφωνία Iceland iSave. Ε, πριν από εβδομάδα υπήρχαν διαπραγματεύσει με τη Ισλανδία και μπορείτε να πείτε ότι στο Λονδίνο και οι Υπουργοί Οικονομικών έχουν δικαίω γιατί πολλοί επένδυσαν στην iSave. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να είμαι σίγουρη ότι οι απαιτήσει προς την Ισλανδία είναι λογικές και αναλογικές. Η Ισλανδία θα πρέπει να είναι καλόδεκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν θα μπορεί να δεχθούν να ταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν στη Υπουργή Οικονομικών, στη Χάγη και στο Λονδίνο τους πιέζουν. Θα πρέπει να δείξουμε μία αλληλεγγύη με την χώρα αυτή. Θα πρέπει να λύσουμε από κοινού τα προβλήματά μας. Και η τελευταία πρόταση στα Ισλατικά. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη. Sir, my information is that you have already... Yeah, there is no, there is no point, point of order. Δεν υπάρχει διαδικαστικό εδώ, σε αυτή τη διευθυνσία. εκτός μικροφώνου παρέμβαση. Personal statements can come at the end, but not, not at le decía, le decía, señor presidente. Σας έλεγα ότι η κυρία Μουνίθε με ναι, αναφέρθηκε σε μένα ρητά, γι' αυτό έχω δικαίωμα ανταπάντησης. Ναι, στο τέλος όμως, όχι τώρα. Thank you. Please. Merci, si θα ήθελα να βάλετε από την αρχή το χρόνο μου στις 28 Φεβρουαρίου γνωρίσαμε την θύελα Ξύνθια η οποία έπληξε τη Γαλλία, ιδιαίτερα τη Δυτική Γαλλία. Σκεφτόμαστε βεβαίως τα θύματα και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τον πληθυσμό. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τους άμεσα θυγόμενους με ένα ταμείο αλληλεγγύης. Πώς τέσσερα με πέντε χιλιάδες άτομα μπορούν να ζουν σε μία πλημμυρισμένη περιοχή. Βλέπουμε ότι ο πρόεδρος Σαρκοζή ζητούσε εδώ και μήνες να υπάρχει ή να δίνεται άδεια κατασκευών σε περιοχές που μπορούν να πλημμυρίσουν, να γνωρίσουν πλημμύρες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια συγχρηματοδότηση υπό τον όρο ότι λαμβάνεται υπόψη η αιγιαλίτιδα ζώνη έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε αλληλέγγυοι σε αυτούς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα, ιδιαίτερα σε αυτούς που, ως προς αυτούς που καλλιεργούν μαλακόστρακα. Ο κύριος Φόξ είναι ο επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. έχει ε, μια παραγωγή στην ε, κρασιού στην ε, εκλογική μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα όμως υπάρχουν ε, επιθέσεις κατά αυτού ε, γιατί οι αισθητικοί θεωρούν ότι το κρασί αυτό φταίει και όχι οι, ε, και πρέπει να καταργηθεί επειδή περιέχει και ε, καφέ και είναι απειματικό και θα γίνει στο μέλλον θα, απογορευτεί το Irish Coffee επειδή έχει και ενόπνευμα και καφέ. Τι κράτος είναι αυτό που μας δαντεύει κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να μπορεί ο καθένας να πίνει ό,τι θέλει και να μην εμπεριφθούν κυρώ στην πλειοψηφία επειδή μερικοί ε, κάνουν καταχράσεις. Και μην νομίζετε ότι αυτοί οι χούλιγαν που πίνουν αυτή τη στιγμή αν απογορευτεί θα πίνουν τσάι. Ευχαριστώ κύριε Φόξ. Κύριε Σταβαρές, ένα λεπτό. Um Ευχαριστώ. Εδώ και ένα χρόνο το ευρώ ήταν δυνατό. Οι οικονομίες όμως του ευρώ είναι διαφορετικές. Γι' αυτό και καταρακώθηκε το ευρώ. Δρούν σήμερα δυστυχώς οι κερδοσκόποι. Κανένας δεν μας υποχρέωσε να προβούμε προς την ΟΝΕ και κανένας δεν μας όρισε να καταφερόμαστε κατά των αδύναμων οικονομιών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για περιφερειακές οικονομίες όπως ονομάζονται. Όμως, τη στιγμή που μιλάμε για ευρώ, θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη και δεν μπορούμε να μιλάμε για περιφερειακές οικονομίες. Αυτό το είδαμε με την επανένωση της Γερμανίας. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη. Ας δράσουμε και εμείς αλληλέγγυα. Obrigado. Thank you. Mr. Agnew. Ευχαριστώ κύριε Σένιο. Κύριε Πρόεδρε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενορμονίσει τα πάντα οδηγεί σε πολλά θύματα, παραδείγματο χάνει και όσον αφορά τα όργανα για την μετεωρολογική καταγραφή των γεγονότων που εξυπηρετούν τους πιλότους του Ηνωμένου Βασίλειου, γιατί υπάρχουν κάποια όργανα που δεν ε, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν, που είναι πραγματικά συγκεκριμένα για το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε πάρα πολύ ομίχλη και άλλα καιρικά φαινόμενα και έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή διαγρα... θέλουν να διαγραφούν και το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί ιδιώτες πιλότοι δεν θα μπορούν να πετάνε εκτός αν υπάρχουν καθαροί ε, καθαροί ουρανοί καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού Γιατί ένας πιλότος έχει 15 δευτερόλεπτα μονάχα για να ξανακερδίσει την ε, σταθερότητα του αεροπλάνου, την έχει χάσει λόγω καιρού. Λοιπόν, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας ε, στον ε, τομέα των μεταφορών να ξανασκεφτεί το θέμα. Εδώ έχουμε πάλι ένα παράδειγμα λογικού νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου που καταγράφεται, που διαγράφεται λόγω της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγγέλικα Βέλμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξότιμοι συνάδελφοι, ένας από τους στόχους της Σχεδιατίας είναι το, η μείωση κατά το ίμιση του διεθνής Το έτος 2010 χαρακτηρίζεται ως το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση ένδυας. 16% των Ευρωπαίων ζουν κάτω από το κατόφλι της ένδυας. Το 79% των Ευρωπαίων ζουν με λιγότερο από το 60% του μέσου όρου εισοδημάτων της χώρας τους. Το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 ε, θα πρέπει να αποδώσει αποτελέσματα στον αφορά την καταπόλυμψη της ε, πτώχειας και του αποκλεισμού. Ευχαριστώ η κυρία Στάρας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρέμβω διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πώς ισχύει ο Ισπανικός νόμος στο ε, νησί Φορμεντέρα που ε, ανήκει στις ε, Βαλεαρίδες νήσους. Η εφαρμογή αυτού του νόμου που ήταν πολύ καλή σε ορισμένες ζώνες δεν μπορεί να ισχύσει στη Φορμεντέρα διότι οι περισσότερες τουριστικές υποδομές από τις οποίες ζει η νήσος που ισχύουν εδώ και 40-50 χρόνια δεν θα υπάρχουν πλέον και το ξενοδοχείο Ροκαμπέγια που ήταν ε, ένα από τα πρώτα της νήσου και ήταν γνωστό διεθνώς και προωθούσε και τη φήμη του νησιού στο εξωτερικό, σύμφωνα με αυτό το νόμο, θα υποστεί μεγάλες αρνητικές συνέπειες. Γι' αυτό θα, θα, θέλαμε να βρεθεί μία διαφορετική λύση για την Φορμεντέρα, έτσι ώστε να τηρείται η ιδιωτική ιδιοκτησία όπως όρισε και το δικαστήριο του Στρασβούρου και να μην ορίζεται ένας νόμος ο οποίος θα ισχύσει αναδρομικά τη στιγμή που οι υποδομές αυτές ίσχυσαν και τήρησαν τις προδιαγραφές εδώ και 30 ή 40 χρόνια. Και αυτό σε σχέση με την Αιγιαλίτιδα ζώνη. Ευχαριστώ. Mr. De Rosa, for one minute. De Rosa, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απάντηση που έλαβε πρόσφατα, πρόσφατα ο Μπούζεκ από τον Νατανιάχου όσον αφορά την είσοδο της αντιπροσωπείας ε, πέρυσι χρειάζεται μια βαριά ανταπόκριση. Στη Γάζα και στην Ιερουσαλήμ δεν μπορεί να απαγορεύει ούτε να παρεμβαίνει με τα δημοκρατικά δικαιώματα αυτού του Ευρωκοινοβουλίου. Η εκπρόσωπος Άνστον θα πρέπει να επισκεφτεί τη Γάζα και θα πρέπει να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει την πολιορκία και την κρίση. Γκόλστον αποκαλεί αυτό παράνομη τιμωρία του πληθυσμού. Χαίρομαι για τη συμφωνία, για συνομιλίες, αλλά κλιμακώνονται οι εντάσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στην Χέμπρον και στην Ευρώνα και θα ήθελα η Άστον να φροντίσει να αποκλιμακωθούν αυτές οι εντάσεις. Ο κύριος Κέλαμα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Όπως μας υπενθύμισε ο Πρόεδρος, στις 11 Μαρτίου η Λιθουανία και η Εσθονία έχουν την 20η επέτειό τους σε σχέση με δύο βασικά νομοθετήματα. Η Λιθουανία κήρυξε την ανεξαρτησία της και στο Ταλίν έγινε η αποκατάσταση του νομικού καθεστώτος το Κογκρέσο της Εστονίας ε, παρουσίασε μια μοναδική εναλλακτική δημοκρατική λύση. Εξελέγει με 90% του πληθυσμού την 30 πολιτικά κόμματα. Στην προσπάθεια λοιπόν αποκατάστασης της πραγματικής ανεξαρτησίας και ενός ε, κράτους ανεξάρτητου προχωρήσανε. Όλα αυτά μπορέσαν όμως να λουποθούν τελικά χάρη στην αλληλεγγύη της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κρέτου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε τόσο καλά ευθυμογραμμισμένοι με όλα που πιστεύω ότι σήμερα θα έπρεπε να ήμασταν πιο γενναιόδοροι με τις γυναίκες. Θα ήθελα να σας μιλήσω για ορισμένες διακρίσεις στην ε, Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Ρουμανία. Στην Κοπενχάγη έγινε μία δήλωση σε σχέση με ε, άρθρα στον τύπο της ε, Δανίας κατά ενός Ρουμάνου και επίσης ένα κοριτσάκι 13 ετών χρειάστηκε να αυτοκτονήσει επειδή του επιτέθηκαν συμμαθήτριές της στο σχολείο. Επίσης, τα τρένα, τα γαλλικά τρένα υπάρχει μία αφίσα η οποία λέει, αναφέρει ότι θα πρέπει οποιοδήποτε πολίτης να αναφέρει στην αστυνομία όταν δει περίεργες κινήσεις, ιδιαίτερα προερχόμενες από Ρουμάνους πολίτες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι επιδεινώνει την κατάσταση ενδοκινοτικά, διότι αυτό αποτελεί το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς να μην γίνονται διακρίσεις κατά ε, ενός έθνους κατά ενός κράτους ευρωπαϊκή Ένωσης. Ευχαριστούμε. One minute. ένα λεπτό. Θα ήθελα να αναφερθώ στην Ατλαντική ε, στρατηγική και τη Βαλτική στρατηγική και τις σχετικές συζητήσεις. Πολλά λέγονται και νομίζω ότι υπάρχει χώρος και για ανάπτυξη. Η στρατηγική 2020 έχει αποσαφηνίσει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει μόνη της και βεβαίως οι χώρες που βρίσκονται στον Ατλαντικό, η Ισλανδία, η ε, Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία μπορούν να βοηθήσουν πολύ με την ηλιακή ενέργεια, την αλληλεία, την ε, αιωλική ενέργεια και θα ήθελα να ζητήσω από την Ισπανική Προεδρία να δώσει προτεραιότητα σε αυτό το θέμα τους επόμενους μήνες. Αν γίνει αυτό, πραγματικά θα έχουν συμβάλει ουσιαστικά ε, μέχρι το τέλος της Προεδρίας τους. Ευχαριστώ, κυρία Πατρόνεβιτς, τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τους τελευταίους τρεις μήνες στην Πορτογαλία ζήσαμε έξι βασικά ε, ναυάγια όπου χάσαν τη ζωή τους 13 ε, αλείς. Χάσαμε ε, πολλά πλοία και τράτες. Στο Ματοζίνιο, σε Τούμπαλ, Αριόζα, Πενής, Καμίνια ζουν ε, αυτά, αυτές οι κομοπόλεις μια κατάσταση πένθους. Ζήσαμε έναν δρυμή χειμώνα και οι αλείς βρίσκονται σε τέτοια επώδυνη θέση που δεν έχουν πόρους ή μέσα. Δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτές τις μηχανότρατες και γι' αυτό ακριβώς ενισχύονται και οι καταστροφές. Αυτό θα πρέπει να εκλείψει. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίζεται η ασφάλεια των αλιέων και αυτό να είναι μία από τις κεφαλίδες των ενασχολήσεων της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, έτσι ώστε οι αλλιείς να έχουν άμεση ε, διασφάλιση, εξασφάλιση των συνθήκων, σωστών συνθήκων εργασίας και της ζωής τους. Υπάρχουν 13 ονόματα στον κατάλογό μου, δεν θα μπορέσω να σας δώσω χρόνο. Ο κύριος Μεσάρος έχει το λόγο και άλλος ένας ομιλητής μόνο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να έχουμε μία σωστή προσέγγιση, ενοποιημένη προσέγγιση της κατάστασης του κοσυφοπεδίου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μία ενία προσέγγιση στην εξωτερική μας πολιτική. Το Κωσυφοπαίδιο αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος από 65 χώρες και 24 χώρες του ΝΑΤΟ, καθώς και 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία να βάλουν στην άκρη τις ανησυχίες τους και να συγκλίνουν με την πλειοψηφία αναγνωρίζοντας το κοσυφοπαίδιο το συντομότερο δυνατόν. Αυτό θα ήταν ένα πολύ σωστό μήνυμα της ολοένα και μεγαλύτερης ενότητας και ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τελευταίος κ. Μπρόντς. Ε, το, κεφαλαίο, το κεφάλαιο κινείται ανά το κόσμο νόμιμα και παράνομα και τα αγαθά και οι υπηρεσίε κινούνται γύρω από τον κόσμο για να μειωθούν οι τιμές και κλείζουν έτσι εργαστήρια, ε, επιχειρήσεις ε, και μένουν πολλοί χωρίς δουλειά και χωρίς χρήματα. Ανοίγονται επιχειρήσεις σε χώρες που υπάρχουν πολύ χαμηλά ημερομίσια Κλείνοντα εδώ στην Ευρώπη. Όπου υπάρχει μια οικονομική κρίση, όλοι οι πολιτικοί εκφράζονται κατά του προστατευτισμού. Μόνο ο προστατευτισμό όμω θα μα επιτρέψει να ξαναδημιουργήσουμε μια επιχειρησιακή βάση και να εξασφαλίσουμε τα μέσα διαβίωση για του ανθρώπου. Η οικονομία είναι προ όφελο των ανθρώπων κανονικά. Δεν είμαστε εμεί υπέρ ε, και προ όφελο των οικονομικών ε, παραγόντων. Βλέπουμε τι συμβαίνει και θα πρέπει να το αποτρέψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σιτρικάκης για μια προσωπική δήλωση σύμφωνα με τον κανόνα 151. Eh, ναι, βασίζομαι στο άρθρο 150. Λυπάμαι που συγχαίρει κάποιος τον Τσάβες, ο οποίος συνεργάζεται με τους τρομοκράτες και την ΕΤΑ, όπως ε, ελέγχθη. Και θα ήθελα να σας πω ότι δεν, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι εμείς δεν θα υποστηρίξουμε τον Θαπατέρο. Δεν μπορείτε να δεχτείτε αυτή τη στάση τη στιγμή που υποστηρίζετε και ο Τσάβες και η διεθνής τρομοκρατία με, τις διμερείς, με τη διμερή αυτή συνάντηση. Ευχαριστώ. Μια καλή διακράτα. Ναι, όσον αφορά τη ζήτηση, τελευταία συζήτηση, θα ήθελα να πω ότι εκφράσαμε την δυσαρέσκειά μας ότι προφανώς δεν είναι σαφές όταν παίρνουμε το λόγο ε, να ξέρουμε πότε περίπου θα μιλήσουμε. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μαθαίνετε από το παρελθόν και δεν προσπαθείτε να διευκολύνετε την ζωή των βουλευτών και να υπάρχει μια ξεκάθαρη διαδικασία. Εδώ και πέντε ε, συνόδους έχω ζητήσει να λάβω το λόγο. Δεν τον έχω λάβει ούτε και σήμερα και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται και πώς παίζει το παιχνίδι. Εγώ ακολουθώ τη διαδικασία. Αλλά θα πρέπει να λάβετε και υπόψη σας ότι έχουμε πάνω από 60 αιτήσει και έχουμε 30 λεπτά για τη διαδικασία αυτή. Και σας έδωσα σε 35 το λόγο. Θα σημειώσω το όνομά σας και θα σας υποσχεθώ ότι την επόμενη φορά θα είστε από τους πρώτους που θα μιλήσετε. Θα ήθελα να σας δώσω σε όλους τους λόγους, αλλά δυστυχώς δεν είναι δυνατόν. Elnök Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να πω ακριβώς τα ίδια όπως ο συνάδελφός μου. Εδώ και έξι μήνες δεν έχω πάρει χρόνο αγόρευσης σε ε, παρεμβάσεις ενός λεπτού. Και θα ήθελα και εγώ να μπορέσω να μιλήσω. Mr. I personally... Κύριε Τέκες, εγώ προσωπικά τουλάχιστον μία φορά σας έδωσα το λόγο. Δεν είναι σωστό να λέτε ότι δεν μιλάτε ποτέ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω. Να δηλώνετε τα ονόματά σας πριν αρχίσουμε. Και θα σας έχουμε στο κατάλογο και θα σας την επόμενη φορά θα σας δώσουμε το λόγο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ τώρα πάρα πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση De Bruyne για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στους μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις